Ε, πρακτικούς τρόπους οργάνωσης ε, των ευρωεκλογών του 2014. Και θα δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Νταφ για να μας παρουσιάσει την έκθεσή του. Έχετε τέσσερα λεπτά κύριε Νταφ. Ε, Πρόεδρε, κυρία Επιτροπέ, παρά το ότι το κοινοβούλιο μας εκλέγεται με άμεση ψηφοφορία εδώ και 35 χρόνια, εξακολουθούμε να θεωρούμε θα κάτι καινούριο. Έχουμε εκτεταμένες νομοθετικές και δημοσιονομικές αρμοδιότητες και ε, αρμοδιότητες ελέγχου, τις οποίες ε, αξιοποιούμε. Αλλά μας κατηγορούν για έλλειψη δημοκρατικής νομιμοποίησης. Τα εθνικά πολιτικά κόμματα και κοινοβούλια είχαν δυσχέρειες ε, προσαρμογής στη δημιουργία ενός αντιπάλου κοινοβουλίου σε ενωσιακό επίπεδο. Τα μέσα τίνουν να ασχολούνται περισσότερο με τα εθνικά κοινοβούλια και όχι με μας τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ελάχιστα λειτουργούν ως μηχανισμοί διεξαγωγής ε, πολιτικών εκστρατιών. Οι υποψήφοι για το Ευρωκοινοβούλιο επιλέγονται από τα εθνικά κόμματα σε εθνικό και όχι ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε δεν θα έπρεπε να μας εκπλήσει το ότι η συμμετοχή στις ευρωεκλογέ φθήνει και έχει οδηγήσει σε ισχυρισμούς από πλευράς πολλών ότι αυτό το μεγάλης διάστασης ε, πείραμα σε διεθνική ή μεταεθνική δημοκρατία έχει αποτύχει. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε ούτω ώστε οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2014 να είναι μια καλύτερη εμπειρία, μεγαλύτερη επιτυχία για τους ψηφοφόρους και τα μέσα. Η Επιτροπή μου και εγώ θεωρούμε ότι μπορούμε να επιτύχουμε κάτι τέτοιο εάν ενισχύσουμε το ρόλο των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων επιλέγοντας υποψηφίους που θα προωθήσουν τα κόμματα και τα εκλογικά προγράμματα των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. που θα κάνουν μια συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ιδέες, πολιτικές, ψήφους και έδρες. κάνοντας ευρύτερα γνωστές τις πολιτικές συζητήσεις που κάνουμε εδώ ως σώμα. Παρουσιάζοντας τις πραγματικές επιλογές για την επιλογή της επόμενης Επιτροπής, για το ρυθμό και είδος ενοποίησης, για το πώς ε, θα δαπανίσει τους πόρους της η Ευρώπη και για το ποια θα είναι η στάση της Ευρώπης στα διεθνή θέματα και βήματα. Γι' αυτό ο νέος πρόεδρος της Επιτροπής που θα εκλέξουμε με απόλυτη πλειοψηφία του σώματος ε, τον Ιούλιο του 2014 θα έχει ε, μία ε, εκτεταμένη δημοκρατική νομιμοποίηση και εντολή. Ευχαριστώ. Λόγω του χρόνου δεν θα χρησιμοποιηθεί η διαδικασία των γαλάζιων καρτών γιατί αλλιώ δεν θα μπορέσουμε να κλείσουμε τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ κύριε Ντάφ για την παρουσίασή σας. Να δώσουμε τώρα μέσω το λόγο στην κυρία Ρέντινγκ, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, για να μας παρουσιάσει την άποψη της Επιτροπής. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αξιότιμο κύριο Άντριου Νταφ για την, όχι μόνο την σημερινή του παρουσίαση, αλλά με την πάροδο το χρόνο του έχει βοηθήσει έτσι ώστε να δημιουργηθεί αυτός ο ευρωπαϊκός χώρος. Ο Άντριου Νταφ έχει απόλυτο δίκιο. Η συμμετοχή των ψηφοφόρων στις ευρωπαϊκές εκλογές έχει μειωθεί σταδιακά από το 62% το 1979 στο 43% το 2009. Αλλά αυτό παρατηρείται όχι μόνο στις ευρωεκλογές, παρατηρείται κατά παρόμοιο τρόπο και σε εθνικές και σε περιφερειακές εκλογές. Πιστεύω λοιπόν ότι αν ξεκινήσουμε να μελετήσουμε το πώς θα βελτιώσουμε τη συμμετοχή στις ευρωεκλογές, αυτό θα βοηθήσει ταυτόχρονα και την βελτίωση της συμμετοχής στις εθνικές και τις περιφερειακές εκλογές. Η Επιτροπή έχει καταβάλει συνεχείς προσπάθειες για την ενθάρρυνση της πολιτικής συμμετοχής και τη βελτίωση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τα δικαιώματα του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμάστε, η πρώτη έκθεση των πολιτών το 2010 ε, με 25 συγκεκριμένες προτάσεις τις οποίες έθεσα επιτάπητος τότε. Τα καλά νέα είναι ότι αυτές οι 25 προτάσεις έχουν υλοποιηθεί ή είναι στη διαδικασία υλοποίησης. Η δεύτερη έκθεση για την πολιτότητα το Μάιο του 2013 έχει εξετάσει τις διάφορες προτάσεις που λάβαμε από τους ίδιους τους πολίτες τον διάλογο που διεξάγουμε στις τα διάφορα κράτη-μέλη ή στις διαβουλεύσεις που ε, κάνουμε μέσω του διαδικτύου είτε ε, λαμβάνοντας ε, την ουσία των, του εκατομμυρίου ετοιμάτων που λαμβάνει η Ένωση κάθε χρόνο. Λοιπόν, θέσαμε και πάλι 12 προτάσεις οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν πριν από το πέρας της ε, θητείας. Μία από αυτές τις προτάσεις είναι για ε, ισχυρότερη ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τα εκλογικά τους δικαιώματα, ιδιαίτερα για αυτούς που ψηφίζουν για πρώτη φορά. Η Κομισιόν θα ε, μετά ε, το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών ε, με την εμπειρία που έχει κερδίσει αυτό το χρόνο θα δημιουργήσει ένα βιβλιάριο με τα κυριότερα ευρωπαϊκά δικαιώματα των πολιτών σε απλή και σαφή γλώσσα. Εκτός αυτού θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε και να αναπτύξουμε τον ευρωπαϊκό δημόσιο χώρο. Αυτό που είδαμε στα ευρωβαρόμετρα, για παράδειγμα, 8 στους 10 πολίτες μας αναφέρουν ότι θα είχαν μεγαλύτερα κίνητρα να ψηφίσουν αν γνώριζαν περισσότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλές φορές υπάρχει ένα έλλειμμα γνώσεων γνώσεων των, δικαιωμάτων, των δυνατοτήτων και του τι ακριβώς κάνει αυτό το σώμα για τους ίδιους τους πολίτες. Ε, πραγματικά έμεινα έκπληκτη ε, στους διαλόγους με τους πολίτες σχετικά με την έλλειψη γνώσης ανάμεσα στους πολίτες για τα αποτελέσματα και τις εξουσίες ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ένα άλλο ευρωβαρόμετρο δείχνει ότι 7 στους 10 πολίτες πιστεύουν ότι εάν γνώριζαν περισσότερα για τα εθνικά κόμματα και την ε, συμμετοχή τους ε, στα ευρωπαϊκά κόμματα, τότε αυτό θα βοηθούσε τα μάλα και 6 στους 10 πιστεύουν ότι αν έχουν ε, υποψήφιους ε, για την ε, Κομισιόν αυτό θα βοηθούσε επίσης την προσέλευσή τους και με βάση αυτό στις 12 Μαρτίου η Κομισιόν εξέδωσε σύσταση στη εθνικά και ευρωπαϊκά πολιτικά ε, κόμματα ε, για την ενίσχυση ε, της διεξαγωγής των ευρωπαϊκών εκλογών με διαφάνεια και συμφωνούμε απόλυτα στις προτάσεις μας με τα λεγόμενα του Άντριου Νταφ. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο και τον εισηγητή συγκεκριμένα που έθιξε όλα αυτά τα θέματα και επίσης που ακολούθησε τις προτάσεις των συστάσεών μας. Ε, συμπίπτουμε και συμπλέουμε στις περισσότερες προτάσεις και κυρίως στην βούληση να ενισχύσουμε την νομιμότητα τη διαδικασία λήψη αποφάσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, τη προσέγγιση αυτού του συστήματο περισσότερο προ του πολίτε. Επίση, αναφέρεται ε, στην ε, ανάγκη μιας ε, εκστρατείας, προεκλογικής εκστρατείας με βάση τα προγράμματα των κομμάτων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα αποστείλει θετικά μηνύματα στους πολίτες σε όλη την Ευρώπη. Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν για τι ψηφίζουν και θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, θα πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκονται οι εκλεγμένοι ψηφοφο... Ε, υποψηφοί τους και τι πρόγραμμα θα ακολουθήσουν. Επίση, η Κομισιόν θέλει να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα ε, των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων, διότι αυτή η πρόταση θα δώσει στα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα μεγαλύτερη ορατότητα και θα του δώσει τη δυνατότητα να λειτουργήσουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντα έτσι μια πραγματική ευρωπαϊκή υπόσταση. Αυτό επίση θα είναι πολύ σημαντικό και ξέρω ότι μπορώ να στηριχθώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να συνεργαστούμε και να πετύχουμε του στόχου μα. Σας ευχαριστούμε κυρία Ρέντινγκ. Περνάμε τώρα στους ομιλητές εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Πρώτα για δύο λεπτά, ο κύριος Σέπφλιν, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Συγχαρητήρια στον κύριο Νταφ, καταρχήν. Ήταν αξιέπαινο το έργο του στο θέμα αυτό. Η έκθεση προσπαθεί να εξασφαλίσει επιτυχή διεξαγωγή των επόμενων ευρωεκλογών. Ταυτόχρονα θέλουμε με την έκθεση να εξασφαλίσουμε στο μέτρο του δυνατού ευρωεκλογέ με ιδιαίτερη έμφαση στο ευρωπαϊκό τους χαρακτήρα. Γιατί μερικές φορές ε, ε, γίνεται μια καπήλευση του χαρακτήρα των εκλογών ε, και παρεκτροπή σε εθνικά συμφέροντα. Μερικές φορές χρησιμοποιούνται βέβαια οι ευρωεκλογέ από τους πολίτες ως ε, ψήφος ε, διαμαρτυρίας και δεν ενδιαφέρονται περισσότερο για αυτά που συμβαίνουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν γνωρίζουν και πολύ καλά τα θέματα οι ψηφοφόροι και η λύση που προτείνει η έκθεση είναι ότι ε, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα μπορούν να έχουν ενισχυμένο ρόλο στις εκλογές και να ορίσουν τους υποψηφίους τους για τη θέση του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η λογική είναι ότι με τον τρόπο αυτό ο επόμενος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα έχει μεγαλύτερη νομιμοποίηση και θα είναι πιο υπόλογος απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό το βήμα, αυτή η εξέλιξη σημαίνει ότι μια πανευρωπαϊκή προεκλογική εκστρατεία θα πρέπει να διεξαχθεί προκειμένου να αφυπνίσει τους Ευρωπαίους πολίτες ε, ως προς τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα της πολιτικής. Γιατί με τον τελευταίο καιρό ένα μεγάλο τμήμα των εξουσιών πέρασε από το εθνικό επίπεδο στο ευρωπαϊκό. Και έτσι οι κοινοτικές αρμοδιότητες επεκτάθηκαν. Η διαδικασία αυτή δείχνει ότι είναι ζωτική σημασία οι ευρωπαϊκές εξουσίες να αιμοποιούνται στο επίπεδο που ασκούνται, δηλαδή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και οι επόμενες ευρωεκλογέ θα έχουν αποφασιστική σημασία προς την κατεύθυνση αυτή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σέπλινγκ. Για δύο λεπτά τώρα και εκ μέρους των σοσιαλιστών το λόγο έχει ο κύριος Ρομπέρτο Γουαλτιέρη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με την ε, εισαγωγή και θέσπιση των άμεσων εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο και μετά με την αύξηση των ε, προνομίων και αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στηρίζεται πια σε μια διπλή νομιμοποίηση, σε αυτή των πολιτών και στην νομιμοποίηση των χωρών. Και με την εξέλιξη αυτή που κυρώνεται και από τη συνθήκη της Λισαβόνας, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υλοποιήσει τους στόχους της, αλλά για κάτι τέτοιο ε, χρειάζεται ένας ευρωπαϊκός δημόσιος χώρος. Με το ψήφισμά μας προτείνουμε πρακτικές προτάσεις που δεν είναι ούτε συνταγματικές ούτε νομοθετικές, αλλά ληφθούν υπόψη θα ενισχυθεί ο ευρωπαϊκός χαρακτήρας των ευρωεκλογών του 2014. Επίσης, ε, επικεντρωνόμαστε στη βασική καινοτομία, στο γεγονός δηλαδή ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα καθορίσουν, θα ορίσουν τους υποψηφίους τους για τη θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό θα τροποποιήσει τη σχέση εμπιστοσύνης ε, μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτή την ιδέα θα πρέπει να την αισθενιστεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί μερικοί όπως η κυρία Μέρκελ φάνηκαν επιφυλακτικοί. Θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως προβλέπει η συνθήκη, εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα πρέπει το Συμβούλιο να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών και να ορίσει τον υποψήφιο μετά από διαβουλεύσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ουσιαστικά θα εκλέξει τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα πρέπει να αναφέρεται λοιπόν μόνο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Επίσης θα πρέπει του χρόνου να ψηφίζουμε για ένα ευρωπαϊκό κόμμα και έτσι ο πολίτης θα ξέρει ποιον υποψήφιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιλέγει. Πρέπει φυσικά όλα αυτά να γίνουν με πολύ εκτενείς προεκλογικές εκστρατείες για να δημιουργήσει και ο ψηφοφόρος εμπεριστατωμένη γνώμη αν υλοποιηθούν οι πρωτοβουλίες της έκθεσης, οι επόμενες ευρωεκλογέ ε, θα είναι ορόσημο και σημείο καμπής ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Σας... Ένα λεπτό για τους φιλελευθέρους, η συνάδελφος Τάιν. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπή, στις επόμενες ευρωεκλογέ τον Μάιο του 2014, λόγω της κρίσης στην Ευρώπη, Περιμένουμε περαιτέρω μείωση της συμμετοχής και πιο ακραία αντιευρωπαϊκά κόμματα. Πώς μπορούμε να σταματήσουμε αυτή την πορεία με τα μέτρα που θα αποφασίσουμε αύριο. Πρώτον, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν στα ψηφοδέλτια τα ονόματα και τα λογότυπα των ευρωπαϊκών κομμάτων, ούτω ώστε να ξέρουν οι εκλογείς ότι αν με εκλέγουν εμένα ως εκπρόσωπο του Γερμανικού Δημοκρατικού Κόμματος εκλέγουν παράλληλα κάποιον από την οικογένεια των φιλελευθέρων. Διότι το όνομα της πολιτικής ομάδας Άλντε είναι σχεδόν άγνωστο στη Γερμανία. Δεύτερον, θα πρέπει έγκαιρα τα πολιτικά κόμματα να ορίσουν τον υποψηφιό τους για την θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία με ευρωπαϊκά θέματα και όχι μέχρι, όπως μέχρι στιγμής με εθνικά θέματα ούτως ώστε μετά τον ε, εκλεγέν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσει για πρώτη φορά με βάση τη στήκη της Λισαβόνας να εκλέξει απευθείας τον ε, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιπλέον. Πρέπει να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες υποψήφοι. Οι γυναίκες είναι η πλειονότητα των Ευρωπαίων και αυτό πρέπει να φαίνεται και στην πολιτική και να θεωρούν και οι γυναίκες ότι εκπροσωπούνται. Ευχαριστώ τον συγητή κύριο Ντάφ για την ε, ευρείας κλίμακας εργασία του και τις ιδέες του ε, για διεθνικά ψηφοδέλτια που μέχρι στιγμής δεν έχουν επιτύχει. 1,5 λεπτό έχει τώρα η συνάδελφος Αντρίν Μπελή από πλευρά των Πρασίνων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ και συγχαίρω τον συγκητή για την εργασία του. Το 2014 θα είναι οι πρώτες ευρωεκλογές μετά την ε, αρχή ισχύω της Συνθήκης Λισαβόνας που αύξησε τις αρμοδιότητες του Λισαβόνα. Αλλά επειδή υπάρχει κρίση εμπιστοσύνη έναντι τη πολιτική γενικότερα και των ευρωπαϊκών θεσμών ειδικότερα, έχουμε ευθύνη να ξαναδώσουμε έννοια και ενδιαφέρον στη διαδικασία καθορισμού των Ευρωβουλευτών. Αυτό είναι ο στόχο τη έκθεση. Να αυξηθεί η διαφάνεια, να αυξηθεί η δημοκρατικότητα και η ευρωπαϊκή διάσταση των εκλογών αυτών. Πρέπει λοιπόν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να έχουν ουσιοδό πολιτικά προγράμματα να παρουσιάσουν υποψηφίου για την ε, θέση του Προέδρου της Επιτροπής το ταχύτερο. Να εκδημοκρατήσουμε και να πολιτικοποιήσουμε τις εκλογές αυτές, να αυξηθεί η συμμετοχή στη διαδικασία αυτή λειτουργία της Ευρώπης. Ο μέλλον πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να προκύψει από αυτό το κοινοβούλιο. Άρα εμέσως από την ψήφο των πολιτών μας πρέπει να εκλεγεί με βάση ένα πρόγραμμα για την Ευρώπη που θα έχει επειρασπιστεί και θα παρουσιάσει σε συζητήσεις ε, με τους άλλους υποψήφου στην Ευρώπη. Αύριο στην ψηφοφορία θα απαιτήσουμε να υπάρξει αυστηρή ισοτιμία ανδρών και γυναικών και να ζητήσουμε προκριματικές εκλογές σε όλα τα κόμματα για το καθορισμό των ε, υποψηφίων τους για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τη θέση του Προέδρου. Ένα ερώτημα τίθεται για το 2014. Το Κοινοβούλιο θα είναι σαν το Συμβούλιο, ένα κοινοβούλιο εθνικών εγωισμών ή θα είναι η έκφραση πολιτικής αναγέννησης μιας Ευρώπης πολύ πιο κοντά στους πολίτες. Αυτό εξαρτάται κυρίως από εμά. Μερικά από τα συστατικά ε, της προσπάθειας αυτής είναι στην έκθεση DAF, είναι ένα βήμα προ μια, προς μια Ευρώπη που θα είναι πιο κοντά στους πολίτες, πιο πολιτική και δημοκρατική. Ευχαριστώ Σαντρίν. Από πλευρά των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, 1,5 λεπτό η κυρία Δεμαρτίνη. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Κύριε Νταφ, καλό είναι να θεωρήσουμε τους κανόνες για τις επόμενες ευρωεκλογέ, αλλά αλλού βρίσκεται το πρόβλημα. Το πρόβλημα βρίσκεται στην αποτυχία του ευρωπαϊκού μοντέλου, ε, που έπρεπε να ευνοεί τους πάντες, ε, αλλά αυτό που συνέβη στην πραγματικότητα είναι ότι το βιωτικό επίπεδο των Ευρωπαίων πολιτών κατακριμνίστηκε. Το 2014 θα είναι μια λιδία λίθος ε, για την ιστορία της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ρομπέρτο Μπερίνη έχει επιλεγεί να εκπροσωπεί στην Ιταλία στα 150, στους για τα 150 χρόνια της Εθνικής Ενότητας. Και δεν θα πρέπει να δοθεί η εντύπωση ότι η Ιταλία είναι μια χώρα που απλώς ε, κατασπαταλάει τους ε, πόρους της. Είναι μια πολύ σφαλμένη εντύπωση και δεν θέλει η Ιταλία να στενέψει ε, από κανέναν για να σωθεί από την κρίση και χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα ε, βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού εξαιτίας μιας ευρωπαϊκής πολιτικής που μέχρι τώρα προστάτευε τις τράπεζες. Η Ιταλία πληρώνει πολύ περισσότερα από ό,τι θα έπρεπε. Είναι ε, βασικός ε, εισφορέας. Γίνεται μια αφέμαξη των Ευρωπαίων πολιτών. Θα πρέπει κάποια στιγμή να πούμε φτάνει πια. Φαίνεται ότι δεν το αντιλαμβάνονται οι κυβερνήσεις που εμένουν στη λιτότητα. Έτσι πριονίζουν το κλαδί στο οποίο κάθονται η Ευρώπη μετά τις ευρωεκλογέ θα πρέπει να γίνει Ευρώπη των Αθηνών και όχι μόνο Ευρώπη των Τραπεζών. Ευχαριστώ. Εκ μέρου τη Ευρώπη για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία για 1,5 λεπτό το λόγο έχει ο κύριο Άγνιου. Well, Νομίζω θα τα πάτε καλά, κύριε Πρόεδρε, διότι νόμιζα ότι είχα μόνο 60 δευτερόλεπτα. Ξεκινάμε και πάλι. Άλλη μια προσπάθεια να στρεβλώσουμε τη δημοκρατία στη Βρετανία. Εάν πραγματικά θέλετε να θέσετε τα εμβλήματα αυτών των πανευρωπαϊκών ομάδων στα ψηφοδέλτια του χρόνου, κάντε το. Κανένα πρόβλημα. Αλλά θα συγχύσετε πλήρω του ψηφοφόρου μα. Σχεδόν κανεί στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει ακούσει από την, για την ECR που είναι μέρο του ονόματο που ονομαζόταν το Συντηρητικό Κόμμα. Ωστόσο, χρησιμοποιώντα αυτά τα παρήεργα ονόματα, είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσετε τα μετρητά των φορολογουμένων για να χρηματοδοτήσετε τις Ε, ε Βέβαια, ε, ο μέσος ψηφοφόρος στη Βρετανία δεν θα έχει ακούσει ποτέ για κάποιον που δεν ονομάζεται τον Μπλερ. Βέβαια, προσπαθήστε να επιτρέψετε τις πολιτικές, τα πολιτικά προγράμματα στα μέντια, αλλά κανένα πολιτικό κόμμα δεν θα θέλει να σχετίζεται με την υπόσκαψη του πολιτικού συστήματός μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθείτε απλά να δημιουργήσετε την ιδέα του Ευρωπαϊκού Δήμου με την ελπίδα ότι τα χρήματα των φορολογουμένων θα σας βοηθήσουν δεν θα το κάνουν αυτό. Ευχαριστούμε κύριε Άγνιο. Για 1,5 λεπτό επίσης το λόγο έχει η κυρία Σενκλέρ. Εκ μέρους των μη γεγραμμένων. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αυτές οι εκλογές ε, είχαν συνεχώς μικρότερη προσέλευση και ε, συνήθως ε, ε, ψηφίζουμε σε εθνικά θέματα. Γι' αυτό το σχέδιο για την Ομοσπονδιακή Ευρώπη δεν έχει την συνένεση του δημοσίου του, κοινού. Δεν σας απασχολούν οι ψηφοφόροι της Ευρώπης. Ο Βρετανικός Πολιτικός τύπο, αναφέρεται επικριτικά, ε, κύριε Νταφ, ε, στην ε, εγχείρημα συμμετοχή στι εκλογέ. Αυτό που δεν κατανοείται είναι ότι ο κόσμος δεν το θέλει αυτό. Παρά την παροχή την έκθεση Μπόλς ότι ο, ο κόσμος πραγματικά δεν το ήθελε. Αναφέρεται ότι οι πολίτες εκπροσωπούνται άμεσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στο Ευρωκοινοβούλιο. Ήδη εκπροσωπούνται από μέλη τα οποία έχουν ψηφίσει. Αλλά η παραδοσιακή άποψη του ε, εκπρόσωπου δεν αρκεί για σας. Ε, δεν είναι αυτό που θέλουμε. Δεν, δεν είναι αυτό που θέλει ο, ο λαός και ο κόσμος. Αυτό που θέλετε είναι να εκπροσωπούνται από ανθρώπους που συμφωνούν με τη δική σας Ομοσπονδιακή Ευρώπη. Αυτή που θέλετε κύριε Νταφ, τι, τι έχει σημασία για σας κύριε Νταφ. Αυτό που θέλουμε είναι ένα δημοψήφισμα για την συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θέλουν οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου. Ευχαριστούμε κύριε Σενκλέρ. Ολοκληρώσαμε τους ομιλητές εκ μέρους των ομάδων και περνάμε στους λοιπούς ομιλητές. Για δύο λεπτά πρώτα το λόγο έχει ο κύριος Τσασκόφσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, υπάρχουν λόγοι για ανησυχία σε όλους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαμηλή προσέλευση εκλογές, ευρωεκλογέ αφισβητούνται και επισκιάζονται από εθνικά συμφέροντα και η νομιμοποίηση ακόμα των θεσμικών οργάνων αφισβητείται. Οι πολίτε δεν έχουν την αίσθηση ότι είναι καλά ενημερωμένοι για την ευρωπαϊκή ολοκληρωσία, ότι έχουν επιρροή στην πολιτική πορεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι για να εξευρωπαίσουμε τι εκλογέ. Γι' αυτό και ζητούμε από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να ορίσουν τους υποψηφίους τους ε, για τη θέση του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και να πραγματοποιήσουν πανευρωπαϊκές ε, προεκλογικές εκστρατείες. Όποιος και κερδίσει, με βάση τις συνθήκες της Λισαβόνας, θα ηγηθεί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση πολιτική εντολή. Και για πρώτη φορά θα έχουμε άμεση σύνδεση της ψήφου του πολίτη με την πορεία που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φαντάζομαι θα εκτιμήσουν τη διαφορά οι Ευρωπαίοι πολίτε και με τον εξευρωπαϊσμό της συζήτηση, έχουμε την ευκαιρία να στείλουμε ένα νέο μήνυμα και να κινητοποιήσουμε τους ψηφοφόρους μας ακόμη και στη, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνονται αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Και εδώ αντιμετωπίζουμε τις πιο σημαντικές προκλήσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περισσότερα εθνικά κοινοβούλια το μισό του χρόνο τον αφιερώνουν σε μεταφράσει των συμφωνιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην ενσωμάτωση των δικών μα αποφάσεων στην εθνική νομοθεσία. Οπότε αν καταφέρουμε να περάσουμε αυτό το μήνυμα προ του Ευρωπαίου πολίτε, ίσω ε, αποκτήσουν και οι ευρωεκλογέ σημασία στα μάτια των Ευρωπαίων πολιτών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή, τον Άνδριο Ντάφ για τι προσπάθειές του και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πούμε οτιδήποτε για τον Άντριο αλλά σε καμία περίπτωση ότι μεροληπτεί ή ότι έχει προκαταλήψεις. Για 1,5 λεπτό το λόγο έχει η κυρία Σιλβίκη Γιόμ. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον Άντριου Ντάφ για το έργο που έχει πραγματοποιήσει. Και είναι πολύ σημαντικά τα θέματα που πραγματεύεται η έκθεση. Καταρχήν, μεγάλη αποχή από τις ευρωεκλογέ, κάτι που δείχνει την αδιαφορία των Ευρωπαίων πολιτών για τα ευρωπαϊκά τεκτενόμενα. Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν την αίσθηση ότι δεν επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές αποφάσεις, ιδιαίτερα σε μια δύσκολη κοινωνική και οικονομική κατάσταση. Οπότε θέλουμε να ανταποκριθούμε στην πρόκληση να συνδέσουμε τους πολίτες στη διαδικασία αυτή. Και ε, Πολλέ είναι οι προτάσει έκθεση. Καλύτερη ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών μέσω τη προεκλογική εκστρατεία. Επίση, το θέμα τη ε, εγγραφή στου εκλογικού καταλόγου που μερικέ φορέ αμελείται. Το θέμα του εξοευρωπαϊσμού των εθνικών προεκλογικών εκστρατείων, με την ε, αναφορά της, ε, των πολιτικών κομμάτων και τη σύνδεσή τους με τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, δυνατότητα ψήφο, εκλέγει και εκλέγει σε άλλη χώρα από αυτή τη καταγωγή και ορισμό του υποψηφίου του, στη θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λυπούμε βέβαια που όλες αυτές οι ωραίες προτάσεις ε, μένουν ακόμη στο επίπεδο των συστάσεων. Θα δούμε αν θα ληφθούν υπόψη και σίγουρα θέλουμε μια δραστήρια προεκλογική εκστρατεία για να επαναφέρουμε την εμπιστοσύνη του Ευρωπαίου πολίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό τώρα το λόγο έχει ο Στογιάννοφ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λοιπόν. Επιτέλους έγινε απόλυτα κατανοητό σε όλους ότι οι προσπάθειες ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να γίνει ένα ομοσπονδιακό κογκρέσο Υπάρχει ένα πρόβλημα με τη διερμηνία. Θα σας παρακαλούσα να ξαναρχίσετε την ομιλία σας. Για να σας ακούσουμε από την αρχή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον κύριο Νταφ για την ταπεινότητα με την οποία βλέπω να συνέταξαν, να συνέταξαν την έκθεσή τους. Ε, φαίνεται ότι καταλάβατε κύριε Νταφ ότι αυτό που χρόνια επιχειρείται να γίνει ένα ομοσπονδιακό κογκρέσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο δεν θα συμβεί. Οι εθνικές δυνάμεις που εκπροσωπούν βλέπουν όμως τι ε, κρύβεται πίσω από την ταπεινότητά σας. Όπως ε, παραδεχθήκατε, η συμμετοχή στις ευρωεκλογέ ε, είναι 11% σε ορισμένε χώρες, σε ορισμένε νέες χώρες το 2004. Γιατί λοιπόν νομίζετε ότι οι πολίτες ε, ε, δεν ενδιαφέρονται. Εντάξει, κάθε τόσο ε, λέτε ότι οι πολίτες πρέπει να συμμετέχουν σε συζητήσεις, αλλά αυτό τι σημαίνει και το να βάλουμε διάφορα λογότυπα στα ψηφοδέλτια που δεν τα έχουν ξαναδεί ποτέ με αυτόν τον τρόπο νομιμοποιείται η Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία δεν ε, συμμετέχουν, δεν απέχουν οι, Ευρωπαϊ... οι πολίτες της Ευρώπης από τις εκλογές γιατί δεν ενδιαφέρονται για το ποιος θα είναι πρόεδρος της Κομισιόν αλλά διότι διαπιστώνουν ότι τους βομβαρδίζουν συνέχεια με κανονισμούς οι οποίοι ε, τους εμποδίζουν στην ελεύθερη καθημερινή και συνήθη ζωή τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε για δύο λεπτά τώρα ο κύριος Καζίνη, πρόεδρος της ε, Επιτροπής ε, Θεσμικών Θεμάτων ε, του Σώματος. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Δεν θα επαναλάβω αυτά που ήδη ελέγχθησαν και τους επένους που απίφθηναν για την έκθεση αυτή ορισμένοι συνάδελφοι, για τους οποίους τους ευχαριστώ. Θα επανέλθω ε, σε αυτά που λέει η έκθεση για το συνέστημα συμμετοχής στην Ευρώπη και τη συμμετοχή στις εκλογές. Ξέρουμε ότι ο καθένας μπορεί να είναι Γάλλος, Άγγλος, να αισθάνεται Γάλλος, Άγγλος κτλ. Αλλά μπορεί με υπερηφάνεια να αισθάνεται και Ευρωπαίος. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η διαδικασία των εκλογών. Το είπαν ήδη ορισμένοι και το επαναλαμβάνω η σημασία της συμμετοχής σε ένα ευρωπαϊκό κόμμα με το λογότυπό του και η σημασία της συμμετοχής στη διαδικασία καθορισμού του υποψηφίου για τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν θα είναι βέβαια στο ψηφοδέλτιο αλλά θα τον έχουν προκαθορίσει τα κόμματα. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Πρέπει λοιπόν τώρα να καθορίσουμε και μια συγκεκριμένη προθεσμία που θα πρέπει να ε, τηρηθεί από όλα τα κράτη-μέλη για τη δημοψή, δημοσίευση των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών. Είναι λεπτομέρεια, αλλά είναι σημαντικό. Και κάτι άλλο. Κάνουμε τις ευρωεκλογέ νωρίτερα, όχι μόνο για λόγους ε, πρακτικούς, αλλά για να επιτρέψουμε επίσης ε, ε, να γίνει αισθητή η λαϊκή κυριαρχία. Δεν θα χρειαστεί να, περιμένουμε, να περιμένουμε μήνες για να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της ψήφου των εκλογέων, όπως το λέει και ο εισηγητής. Να καταλάβουν λοιπόν οι εκλογείς ότι μετράει η του. τους. Βεβαίως γίνεται μεγάλη συζήτηση για τις σχέσεις μεταξύ ευρωπαϊκής και ε, εθνικής κυριαρχίας ευρωπαϊκών και εθνικών κοινοβουλίων. Αλλά θέλουμε η κυριαρχία αυτή να είναι κάτι που το καταλαβαίνει ο κάθε πολίτης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Κάρλο. 1,5 λεπτό τώρα. Η κυρία Τζίτα Γκουρμάε. Ευχαριστώ. Γνωρίζουμε όλοι το διακύβευμα των επόμενων ευρωπαϊκών εκλογών. Μια από τι μεγαλύτερε προκλήσει είναι να διασφαλίσουμε ένα γενικό διάλογο. Μπορεί να διαφωνούμε πολιτικά, αλλά είμαι βέβαια ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι οι ευρωπαϊκοί, ευρωπαίοι πολίτε αξίζουν μια εξαρτία που να καθορίζει τι κοινέ προκλήσει που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και ε, τις διαφορετικές πολιτικές εναλλακτικέ. Πρέπει να τονίσουμε και τη διαφάνεια και την ε, δημοκρατική νομιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ε, έχει υποστεί ένα μεγάλο πλήγμα μέσα στην κρίση. Ως εκπρόσωποι των πολιτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε να διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα γιατί το Ευρωκοινοβούλιο έχει εκτεταμένες εξουσίες μέσα από την συνθήκη της Λισαβόνας ως υποψήφοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, προσπίζουμε τα διαφορετικά πολιτικά προγράμματα ε, ε, προσδιορίζοντας τον υποψήφιο για τις κρίσιμες θέσεις όπως φαίνεται και στην συνθήκη της Λισαβόνας. Υποστηρίζω πλήρως τους όρους της εκθέσης και ελπίζω να γίνουν οι σωστές διευθετήσεις έτσι ώστε να ενισχυθεί ο δημοκρατικός βίος των Ευρωπαίων πολίτων. Θέλουμε που να αντιπροσωπεύουν όλη την ε, κοινωνία, γυναίκες, ε, νέους ε, στα ψηφοδέλτια. Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες δεν έχουμε ακόμα ίση εκπροσώπηση, αλλά είναι θέμα δημοκρατίας το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να γείται με το παράδειγμά του και ως ισχυώδης εισηγήτρια υποστηρίζω πλήρως την Βιβιάν Ρντίνγκ. Ελπίζουμε ότι θα πετύχει η λιθανική Προεδρία στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Γκουρμάη και τελευταίος ομιλητής ε, ο κύριος Παύλο Ρανζέλ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω καταρχήν ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο ως ε, μέλος της Επιτροπής Σταγματικών Υποθέσεων που ο Άνδριο Ντάφ ε, κατόρθωσε να φτάσει στο αποτέλεσμα αυτό. Αλλά θα ήθελα να πω και κάτι προς συναδέλφους Νταφ, Γουαλτιέρη και Τσασκόφσκι που έφυγε στο μεταξύ. Χρειάστηκαν μεγάλες πιέσεις για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Χρειάστηκαν πολλές ε, τροπολογίες στην έκθεση για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που φτάσαμε σήμερα. Και χαίρομαι ιδιαίτερως γιατί ήταν πραγματικά τεράστιες οι ε, προσπάθειες και διαπίστωσα απροθυμίες ε, και από κάποιους που είχαν διαφορετική άποψη στην αρχή για τις ευρωεκλογέ του 2014. Χρειάστηκε να πιέσουμε και την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, για να αισθενιστεί αυτή την ε, άποψη που πρεσβεύουμε στην έκθεση. Επίσης, ε, να επιστήσω την προσοχή σε ορισμένα θέματα. Αναφέρθηκε εδώ ότι όλα αυτά δεν έχουν νόημα, οι συστάσεις δεν έχουν νόημα και ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν γνωρίζουν τα αρχικά των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Αλλά αν ε, δεν γίνει η συζήτηση αυτή, η δημόσια συζήτηση, θα μείνουν στην αγνοιά τους. Πρέπει πρώτα να γίνει ευρεία συζήτηση για να γνωστοποιήσουμε στους πολίτες αυτά τα θέματα. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε πρώτα να τονίσουμε τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα των ευρωεκλογών. Αν δεν ε, επιμείνουμε σε αυτή την προσπάθεια, δεν θα αντιληφθούν την κατάσταση αυτοί οι Ευρωπαίοι πολίτες. Γι' αυτό θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο θέμα αυτό. Επίση, ένα επίμαχο θέμα, τον διορισμό υποψηφίου για τη θέση του Πρόεδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί εδώ ε, αυτό το θέμα ε, αφορά μια πολιτική δυναμική και όχι μια νομική και προϋποθέτει ε, μια πραγματική ευρωπαϊκή συζήτηση και ένα πραγματικά ευρωπαϊκό δημόσιο χώρο. Γι' αυτό και ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους για τις προσπάθειες που κατέβαλα και για το αποτέλεσμα που επιτύχαμε στην έκθεση DAF. Ευχαριστώ. Και τώρα περνάμε στη διαδικασία CatchDI. Δεν είναι πολύ. Ένα λεπτό καθένας. Πρώτος ο κύριος Ταραμπέλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία παρέθεση. Κυρία Ντεμαρτίνη, κυρία Ντεμαρτίνη, δεν είμαι σίγουρος ότι ο Ρομπέρτο Μπενίνη δίνει κακή εντύπωση για την Ιταλία γιατί νομίζω ότι πολύ περισσότερη κακή εντύπωση για την Ιταλία δίνει ο πρόεδρος Μπερλουσκόνη με την ε, σύγχυση των, ε, της, των επαγγελματικών και των πολιτικών του καθηκόντων. Θέλω να συγχαρώ τον Άντριο Νταφ ε, για την πρότασή του. Έχουμε ένα πρόβλημα στην εικόνα μας, αλλά φταίμε και εμείς σε μεγάλο βαθμό. Και έχουμε ένα έλλειμμα και επικοινωνιακό. Επίσης, οι ευρωσκεπτικιστές που χαίρονται με την οικονομική κρίση ουσιαστικά είναι αντιευρωπαίοι. Ο κύριος Φαράζ φροντίζει να αποφύγει την καταβολή φόρου στη χώρα του και μεταφέρει τα χρήματά του σε offshore λογαριασμούς. Και έτσι αυτοί οι, ευρώφοβοι και ευρωσκεφτικιστές μας τριμώχνουν και πιστεύω ότι θα πρέπει... Διακόπτει δυστυχώς ο πρόεδρος στο μικρόφωνο του κύριου Ταραμπέλα. Ο κύριος, ο Ευχαριστώ. Δημοκρατία πρέπει να υπάρχει για όλους τους τομείς πολιτικής. Δεν είναι αντικείμενα, αλλά υποκείμενα της πολιτικής οι πολίτες. Όλων των πολιτικών αποφάσεων. Αυτό πρέπει να το διαπιστώσουν οι πολίτες. Και ιδιαίτερα στην Ευρώπη μας. Τι γίνεται σήμερα όταν ε, έχουμε ευρωεκλογές. πολλά κόμματα δεν μιλάνε καθόλου για ευρωπαϊκά θέματα, αλλά για εθνικά. Και όταν περνάνε οι εκλογές, τότε ξεπροβάλλει ένας πρόεδρος επιτροπής που δεν είχε συζητηθεί καθόλου ε, κατά την προεκλογική περίοδο και που τον εξέλεξαν κάποιοι σε κάποιο σκοτεινό δωμάτιο. Δεν είναι τρόπο αυτό για να αυξηθεί η συμμετοχή. Γι' αυτό στηρίζω την πρόταση στο μέλλον τα πολιτικά κόμματα πριν τι εκλογέ να δηλώνουν ποιο θα είναι ο υποψήφιό του για τη θέση Προέδρου τη Επιτροπή και μετά να μπορούν να εκλεγούν μόνο όσοι ήσαν υποψήφοι ακριβώς, είχαν καθοριστεί και φυσικά να από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Κάμπελ Μπάνερμαν τώρα. Κάμπελ Μπάνερμαν. Ο κύριος. Ευχαριστώ. Ξέρω ότι ο κύριος Νταφ είναι αξιεπένος, ε, ε ότι είναι φεντεραλιστής και ότι θέλει ένα ευρωπαϊκό υπερκράτος. Αλλά αυτό υπάρχουν εκατομμύρια πολίτες στην περιοχή μου ε, δεν το θέλουν στην νοτιοανατολική Αγγλία και γι' αυτό δεν υποστηρίζουν ορισμένοι το κόμμα του γιατί δεν είναι υπέρ ε, του δημοψηφίσματος για την συμμετοχή που θα γίνει την Παρασκευή στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Αλλά ακόμη και με τα κριτήρια αυτά, αυτά που λέει για τα εμβλήματα και τις δικές τους ε, ε, τα δικά τους πολιτικά μηνύματα στις ε, τηλεοράσεις είναι απαράδεκτα. Ξέρω ότι το ΕΛΚ ε, ήδη έχει αποφασίσει τον προπολογισμό του. Πολλών εκατομμυρίων είναι γι' αυτό. Τα ευρωπαϊκά ε, πολιτικά κόμματα πρέπει να ορίζουν και τους υποψηφίου τους για τη θέση του Πρόεδρου της Επιτροπής. Αυτή είναι μια προσπάθεια που δεν θα οδηγήσει πουθενά. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε, ο Πρόεδρος. Ο κύριος Ζουάου Φεραίρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φαίνεται ότι επιχειρείται μια διαδικασία μυθοποίησης και εξειδανίκευσης που θα προσπαθήσει να μετατρέψει τις ευρωεκλογές σε κάτι που δεν είναι ούτε μπορούν να γίνουν. Θέλουμε να αποσπάσουμε την προσοχή μας από ένα κεντρικό θέμα των εκλογών, δηλαδή να μην εξετάσουμε τον αντίκτυπο των ευρωπαϊκών πολιτικών σε κάθε χώρα και λαό και τη θέση του κάθε κόμματος σε ό,τι φάρει διαμόρφωση αυτών των πολιτικών και εξέταση εναλλακτικών προτάσεων. Η υπεύθυνοι για την οικονομική ύφεση, τη φτώχεια και την κοινωνική κατακρίνηση θέλουν να μετατρέψουν τις επόμενες ευρωεκλογές σε κάτι διαφορετικό. Σε συζήτηση για τον υποψήφιο το, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τα πολιτικά κόμματα που είναι μακριά από την καθημερινότητα των πολιτών και θέλει να μη λάβει υπόψη την αφαίρεση της κυριαρχίας από το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Και πάλι διακόπτει ο Πρόεδρος. Το λόγο έχει η κυρία Ντότς, τελευταία μιλήτρια στο Catch Ευχαριστώ. Κύριε Νταφ, ε, είστε επίμονος με τα φεντεραλιστικά σας ε, όνειρα. Πιστεύω ότι αυτό γίνεται κατά της θέλησης του Βρετανικού λαού. Δύο-τρεις φορές ήδη ε, έχω σχολιάσει ε, διάφορες άλλες δικές σας εκθέσεις ε, ιδίου φυράματος. Ένας συνάδελφος σήμερα το απόγευμα είπε ότι αυτές οι συστάσεις θα δώσουν νέα ζωή στην Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που μπορεί να δώσει νέα ζωή στην Ευρωπαϊκή Δημοκρατία και την συζήτηση για την Ευρώπη στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι δημοψήφισμα για το εάν θα συνεχίσουμε να είμαστε εντός της Ένωσης. Αυτό το δημοψήφισμα το κόμμα σας κύριε Ντάφ εξακολουθεί να το αρνείτε στο λαό του Ηνωμένου Βασιλείου. Αλλά θα αποφασιστεί την Παρασκευή τέτοιο δημοψήφισμα από το κοινοβούλιο μας. Ελπίζω να σας κάνει να σκεφτείτε αυτό, να καταλάβετε τι σημαίνουν όλα αυτά. Ευχαριστώ κυρία Ντόντ. Τελευταίος ομιλητής ο κύριος Γιάννος Σέμπρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Ντάφ και να, διαψε... και να ε, υποστηρίξω όλους αυτούς που δικαίως είπαν ότι ε, στην προεκλογική εκστρατεία θα πρέπει να προτείνουμε και υποψηφίους μας ε, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί έτσι θα έχουμε καλύτερη ευκαιρία για συζήτηση των ευρωπαϊκών θεμάτων και δεν θα επικεντρωθούμε στην συζήτηση των εθνικών θεμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βέβαια αυτή είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά θα πρέπει να ξεχνάμε και τη θέση των διαφόρων κρατών μελών, ιδιαίτερα τις θέσεις των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων αυτών των χωρών. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Επίτροπο, που είναι υπέρ τη πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η θέση των μεμονωμένων κυβερνήσεων, ώστε να μην ε, καταλήγουμε εμείς σε δίκαια κατά τη γνώμη μας αποτελέσματα, αλλά μετά να μας μπλοκάρει το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τελείωσε ο γύρος της διαδικασίας προσέλκυσης της προσοχής του Προέδρου. Το λόγο έχει η κυρία Βιάννα την αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να αντιδράσει στις παρεμβάσεις ε, που ακούστηκαν. Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για την έκθεση αυτή. Να ευχαριστήσω κυρίως τον εισηγητή για το υπέροχο έργο που έχει κάνει μαζί με τους συναδέλφους του στην Επιτροπή. Αυτή η έκθεση μαζί με τις συστάσεις της Κομισιόν πάνε προς την ίδια κατεύθυνση, δηλαδή προς βελτίωση της ε, προσέλευσης των ψηφοφόρων στις ευρωπαϊκές εκλογές και θα χρειαστεί μια κοινή προσπάθεια και από τα ευρωπαϊκά και από τα εθνικά πολιτικά κόμματα και τα κράτη-μέλη ό,τι μπορεί να κάνει η Κομισιόν θα κάνει ε, για να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Επίτροπε. Και τελευταίος ε, θα ξαναλάβει το λόγο ο εισηγητής μας ο κύριος Νταφ. Ε, έγιναν πολλές εικασίες, ιδιαίτερα για το δικαίωμα και για το τι ακριβώς θέλω να πετύχω. Θα σας πω ακριβώς τι θέλω. Θέλω ένα ισχυρό πλουραλιστικό κοινοβούλιο, όπου οι εθνικιστές και οι αυτοί που είναι υπέρ της Ομοσπονδίας ε, προσωπούνται σαφώς με δημοκρατικό τρόπο. Έχουν αναφερθεί θέματα ότι η οικονομική και χρηματοπιστική κρίση θα μειώσει την προσέλευση περισσότερο. Πρέπει να πω ότι διαφωνώ με αυτό. Σίγουρα, αν ε, καταγόμουν από μια χώρα που υπαγόταν σε πρόγραμμα της Τρόικας, θα ε, πήγαινα από το πρωί να ψηφίσω πρώτος-πρώτος. Και ε, υποψιάζουμε ότι αυτό που πρέπει να κάνουν τα πολιτικά κόμματα είναι να ε, βρουν ε, μια λύση εξόδου από αυτή την βαθιά οικονομική κρίση. Αντιλαμβάνομαι από αυτά που άκουσα ότι δεν είναι τόσο απλό για τα πολιτικά κόμματα να βρουν και να επιλέξουν και να ε, διατηρήσουν υποψήφιου για την Κομισιόν. Ναι, ναι, είναι ένα πείραμα και όλα τα πολιτικά κόμματα θα προσεγγίσουν αυτή την πρόκληση από διαφορετικές πλευρές. Οι πράσινοι έχουν πρώτη τις εκλογές καλή του τύχη. Αλλά είμαι βέβαιος ότι αυτό το πείραμα θα ε, μεταμορφώσει την ποιότητα της ε, εξατία, θα την κάνει πιο εξατομικευμένη, ε, πιο θεαματική αν θέλετε και θα έχει ως αποτέλεσμα ένα ισχυρότερο, ε, πιο διαφανές και πιο νόμιμο πολιτικό σύστημα σε επίπεδο ομοσπονδιακό. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο το μεσημέρι. Περνάμε τώρα στην επόμενη έκθεση. Την έκθεση κυρίας Χολμάιερ για τις επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών. Το λόγο έχει η εισηγήτρια, η κυρία Μόνικα Χολμάιερ. Για τέσσερα λεπτά.